και επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας στον Τάραντα τον Ιούλιο, που πραγματοποιήθηκε 13 και 14 Ιουλίου. Κύριε Μαριά, μπορούμε παρακαλώ να συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα, διότι ο κύριος Λαβία βιάζεται και θα πρέπει να αποχωρήσει σύντομα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να του δώσω το λόγο και μετά θα επανέλθω σε εσά εάν συμφωνείτε. Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με τη διαδικασία Κυρία Πρόεδρε, σύμφωνα με τη διαδικασία πρέπει να ανακοινώσετε τις αποφάσεις των συντονιστών όπου εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με την αναφορά για τις γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις. Επομένως, πρέπει να ανακοινώσετε την απόφασή σας και σας έχω ζητήσει το λόγο επί του θέματος αυτού. Και νομίζω ότι αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Βεβαίω, αν εσείς θέλετε να ακολουθήσετε άλλη διαδικασία, εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω, αλλά η διαδικασία η ορθή είναι να μας ανακοινώσετε τις αποφάσεις, να τεθούν τα ζητήματα εδώ και βεβαίω σας έχω ζητήσει το λόγο επί αντιρρήσεων επί των αποφάσεων που πήρατε για το θέμα των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου στην αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Ευχαριστώ. I would recommend you, Mr. Κύριε Μαριά, προτείνω να διαβάσετε προσεκτικά την ημερήσια διάταξη. Αναφέρεται σαφώς ότι η ανακοίνωση των ε, της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές ε, θα γίνουν στις 3 σήμερα το απόγευμα. Βρίσκονται στη ημερήσια διάταξη εδώ και μήνες στο σημείο αυτό. Τώρα λοιπόν ε, σας δίνω το λόγο, Τζοβάνι. Και όπως ε, ξέρεις θα κάνουμε μια διαρευνητική επίσκεψη στον Τάραντα δεν έχουμε στόχο λοιπόν να ξαναεφεύρουμε τον τροχό. Βρέθηκες εκεί ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχεις να μας πεις και για να προετοιμαστούμε και για τη δική μας επίσκεψη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσω εδώ στην Επιτροπή Αναφορών τα όσα κάναμε ως Επιτροπή ΕΝΒΗ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στον Τάραντα. Η διάσκεψη των Προέδρων ε, ενέκρινε το αίτημα της Επιτροπής μας να στείλει αντιπροσωπεία πρώτα στη Ρώμη και μετά στον Τάραντα για να επισκεφτούμε την βιομηχανική εγκατάσταση ε, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Η πρώτη συνάντηση έγινε στη Ρώμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας ε, του Εδάφους και της Θάλασσας με τον ε, Υπουργό και κάποια ανώτερα στελέχη του προσωπικού του. Πριν και μετά την επίσκεψη στην βιομηχανική εγκατάσταση Ριβαστήλ, ε, συναντηθήκαμε με τοπικές αρχές, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους κύκλους συμφερόντων. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα βασικά αποτελέσματα των συναντήσεων που είχαμε κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπείας μας ε, και να σας πω τι λάθη κάναμε για να σας δώσουμε την ευκαιρία να μην κάνετε τα ίδια λάθη, διότι είναι δύσκολο να καταλάβουν εκεί γιατί υπάρχουν ε, διάφορες αντιπροσωπείες από τον ίδιο φορέα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κάνουν την ίδια δουλειά. Ε, θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να οργανώσετε πρόσθετες ε, συναντήσεις και να υποβάλλετε πρόσθετα αιτήματα για να μπορέσουν να απαντήσουν οι τοπικές αρχές και στους αναφέροντες. Κατά την πρώτη μας συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ε, στη Ρώμη. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό και το προσωπικό του. Καταλάβαμε λοιπόν ε, την μακρά διαδικασία και τις εντολές ε, προς ε, τη βιομηχανία για μείωση της ρήπανσης και για να είναι ε, πιο καλύτερη η ποιότητα ζωής γύρω από την εγκατάσταση αυτή. Το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στην πόλη. Και γύρω από μια τέτοια εγκατάσταση όπως ε, στην Ήλβα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει σαφής διαχωρισμός ε, της βιομηχανικής εγκατάστασης από την πόλη. απαιτείται μία τεράστια περιοχή, ένα χιλιόμετρο επί μισό χιλιόμετρο, όπου ε, υπάρχουν οι πρώτες ύλες που είναι στιβαγμένες ε, σε ύψος 80 μέτρων. και έτσι έχουμε μια τεράστια έκταση η οποία θα πρέπει να καλυφθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και επίσης, όταν φυσάει, ο άνεμος μεταφέρει μικροσωματίδια στην πόλη. Έτσι λοιπόν είναι σαφές ότι θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες η βιομηχανική μονάδα για να καλύψει την πρώτη ύλη για να αποφευθεί αυτό. Εμείς επισκεφτήκαμε τον Ιούλιο την ε, περιοχή αυτή που είναι ιδιαίτερα ξηρή ε, στην Νότια Ευρώπη. Έτσι λοιπόν απαιτείται πολύ νερό που ε, να ψεκάζεται, να καταβρέχουν δηλαδή τις πρώτες ύλες για να αποφύγει για να αποφευχθεί η μεταφορά σκόνης και σωματιδίων στην πόλη. Αλλά οι τοπικές αρχές είπαν ότι θα πρέπει να καλύπτονται οι πρώτες ύλες κάτι που στοιχίζει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν είναι πολύ εύκολο να κατασκευαστεί αυτό το κάλυμα, διότι καταλαβαίνετε ότι διότι πώς θα κατασκευαστεί ένα κάλυμα για μια έκταση ε, ενός χιλιόμετρου επί μισό χιλιόμετρο ε, χωρίς ε, να μπορούν να κατασκευαστούν πυλώνες. Η βιομηχανική μονάδα θέλει να προσφύγει κατά της εντολής αυτής, ε, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία. Αυτή ήταν η πρώτη μας επίσκεψη στη Ρώμη. Μετά καταφτάσαμε στον Τάραντα, συναντηθήκαμε με τον Νομάρχη, με τον ε, Δήμαρχο. Και είχαμε και μια τεχνική συνάντηση με την Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνάντηση αυτή, διότι μας έδωσαν στοιχεία σχετικά με ε, την ε, υγεία των κατοίκων της περιοχής, σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών ε, στην βιομηχανική εγκατάσταση, καθώς και για το τι θεωρούν απαραίτητο να γίνει. Επίσης είχαμε συνάντηση με τις τοπικές αρχές υγείας στον Τάραντα, ενώ αργότερα Είχαμε συνάντηση με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Φυσικά ακούσαμε πολλές διαφορετικές απόψεις. Διότι δεν ήταν πολύ σαφές πώς είναι δυνατόν να συσχετιστεί ε, να συσχετιστούν οι μέρες με ισχυρό άνεμο με προβλήματα υγείας. Ε, τις ημέρες που πνέει ισχυρός άνεμος ε, μεταφέρονται πολλά σωματίδια και έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα υγείας στους ανθρώπους που μένουν κοντά. Ο αρμόδιος ε, για τη λειτουργία της βιομηχανικής εγκατάστασης ε, προσπαθεί να μειώσει τον θόρυβο και τα άλλα προβλήματα. Αλλά απαιτείται πολλή δουλειά για κάτι τέτοιο. Συναντηθήκαμε και με διάφορες ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ακούσαμε τα περί ανεργίας στην περιοχή. και είναι σαφές ότι υπάρχουν προβλήματα. Διαπιστώσαμε καταρχάς το μέγεθος ε, αυτής της εγκατάστασης ε, που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το μέγεθος ε, όντας απ' έξω. Όταν μπει μέσα, συνειδητοποιεί τις αποστάσεις. Συνειδητοποιεί πόσο μεγάλο είναι το απόθεμα των ε, πρώτων υλών. και έτσι μόνο μπορεί να διαπιστώσει κανείς πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι η εγκατάσταση αυτή και ε, οι πόλοι βρίσκονται πολύ κοντά. 100 μέτρα δηλαδή από εκεί όπου αποθηκεύονται οι πρώτες ύλε μέχρι την πρώτη κατοικία. Και είναι σαφές ότι δεν μπορεί κανείς να χτίσει τείχος. Θα πρέπει να μειώσει κανείς ε, την ρήπανση και θα πρέπει να κοιτάξει και την, ε, τις αποστάσεις προς την πόλη. Δεν μπορεί κανείς να βάλει ε, ένα σχολείο δίπλα. Απ' την άλλη δεν μπορεί και να το κλείσει τη στιγμή που εργάζονται 10.000 άνθρωποι εκεί, ιδιαίτερα όχι με τα παρόντα επίπεδα ανεργίας. Γι' αυτό λοιπόν ήταν ε, χρήσιμη η επίσκεψη. Ο ε, αρμόδιος ε, κρατικός υπάλληλος που είναι αρμόδιος μας έδειξε από πού προέρχονται οι πρώτες ύλες. Επισκεφθήκαμε και το λιμάνι, διότι ο μισός λιμένας του Τάραντα ε, το μισό του λιμανιού του Τάραντα ε, ε, προορίζεται αποκλειστικά για τις μεταφορές πρώτων υλών προς την εγκατάσταση αυτή. Έχουμε ε, κυλιόμενους σημάντες. Μήκους 10, 20, 30 χιλιόμετρων για τη μεταφορά των πρώτων υλών. που ε, εν μέρη είναι καλυμμένοι, εν μέρη είναι ε, ανοιχτοί. Περνούν τον αυτοκινητόδρομο, περνούν από διάφορους δρόμους ε, για τη μεταφορά πρώτων υλών από το λιμάνι στην βιομηχανική εγκατάσταση. Και φτάνουν στο σημείο όπου αποθηκεύονται οι πρώτε Υπάρχουν όμως και σοβαρά προβλήματα με τη δικαιοσύνη, διότι, για παράδειγμα, πρέπει να μειωθεί η μεταφορά σωματιδίων όταν καταφτάνει ένα μεγάλο πλοίο και αρχίζει το, η εκφόρτωση των πρώτων υλών. Και αυτό είναι δύσκολο, διότι το λιμάνι βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δικαστικών αρχών ε, λόγω ενός ατυχήματος που πραγματοποιήθηκε το 2010. Έτσι λοιπόν έχει κλειστεί μέρος του λιμένα Έχουν λοιπόν ε, τα υλικά για την μείωση της ρήπανσης, είναι διατεθειμένοι να κάνουν τη δουλειά που απαιτείται, το Υπουργείο τους το ζήτησε αυτό, αλλά δεν μπορούν να εργαστούν στο σημείο αυτό, διότι ε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό τον έλεγχο των δικαστικών αρχών το μέρος του, λιμάν, ε, μέρος του λιμένα λόγω του ατυχήματος που συνέβη. Τέλος είχαμε μία συνάντηση με τον εκπρόσωπο της περιφέρειας της Απουλίας, τον κύριο Εμιλιάνο, που είναι υπεύθυνο ε, για την περιφέρεια, όπως είπα, και Βεβαίω κατανοήσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερη σχέση ανάμεσα στην περιφερειακή διοίκηση και τους αρμόδιους τη ε, βιομηχανία της βιομηχανίας και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διότι πρέπει να συνεργαστούν καλύτερα ώστε να περιορίσουν τη ρήπανση, να μπορούν να, να δουλέψουν σε ταχύτερους ρυθμούς, να μειώσουν το χρόνο που χρειάζεται για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος. Εν τέλει καταλήξαμε ε, ότι Ε, καταλήξαμε μάλλον σε μια συνέντευξη τύπου στο τέλος της επίσκεψης. Αλλά πρέπει να πούμε ότι παρά τις βελτιώσεις που έχουν γίνει, πλήρης σεβασμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ακόμα δεν υπάρχει. Και μάλιστα ε, πρέπει ακόμα να γίνουν πάρα πολλά. Το μέγεθος των εγκαταστάσεων και των παρεμβάσεων που απαιτούνται είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, καθιστούν δύσκολη μάλλον τη γρήγορη ε, διόρθωση όλων αυτών των προβλημάτων. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν χρειαζόμαστε χρόνο για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για το περιβάλλον και ξέρουμε πολύ καλά ότι για την πλήρη συμμόρφωση προς την ε, περιβαλλοντική νομοθεσία των εγκαταστάσεων της ΣΥΛΕΒΑ χρειαζόμαστε σήμερα πάρα πολύ δουλειά. Ε, είναι σαφές ε, ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε το εργοστάσιο αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί η ρήπανση στην περιοχή με πολύ ισχυρές επεμβάσεις και αν χρειαστεί θα πρέπει και να μειώσει η παραγωγή για τη διάρκεια των έργων. Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Είδαμε πόσο η δουλειά έχει γίνει, είναι καλή, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα και όσο γίνεται και πιο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπεριστατωμένη σας παρουσίαση. Η Ιταλία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα χώρα σε, από όλε τι πλευρέ και η Επιτροπή μα, όπω γνωρίζετε, θα επισκεφθεί από τι 2 στι 4 Νοεμβρίου την περιοχή, μια αντιπροσωπεία που θα αποτελείται από 7 μέλη. Εγώ δυστυχώ δεν θα έχω τη χαρά και τη δυνατότητα να πάω εγώ ίδια ότι θα προεδρεύσει την επιτροπή μας εκεί, την αποστολή και ο Εντουάρ Μαρτά. Έχετε και μια έκθεση νομίζω συντάξει για αυτό το θέμα και ίσως λοιπόν πριν από την δική μας επίσκεψη θα μπορούσαν οι γραμματείες μας να δουλέψουν μαζί για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε καλύτερα. Ο κόσμος δηλαδή υποφέρει από το θόρυβο, τη σκόνη, τη ρήπανση εκεί και πρέπει ε, λοιπόν να το δούμε αυτό πάρα πολύ προσεκτικά γιατί είμαστε ο μόνος θεσμός που έχουμε άμεση επαφή με τους δεμονομένους πολίτες. Και τώρα θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Επιτροπής, τον Γιώνα Καμπέσκο, που είναι παρόν. Ε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι σε αυτή την υπόθεση έχουμε ξεκινήσει διαδικασία κατά παράβαση και ότι τα βασικά στοιχεία είναι ότι σε αυτή την περίπτωση οι εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στις άδειες που έχουν πάρει. Ε, ο κύριος Λαβία το ανέφερε, είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, διότι χρειάζονται πάρα πολλοί πόροι, πολλά χρήματα ε, οι εγκαταστάσεις είναι τεράστιες και δυστυχώς ε, όταν έπρεπε δεν έγιναν οι απαραίτητες επενδύσεις. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν που έχει αρκετά προχωρήσει ε, το παρακολουθούν πολύ στενά, αλλά αυτή είναι μόνο η μία πτυχή, είναι η περιβαλλοντική και έχουμε και άλλη μία πτυχή που είναι οι κρατικέ ενισχύσει. Το θέμα είναι λοιπόν ότι σύμφωνα με τους ε, κανόνε περί κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν, ισχύουν για τον τομέα του χάλιβα, τη παραγωγή χάλιβα, δεν είναι δυνατόν το Ιταλικό κράτο να πληρώσει για τέτοιου είδους επενδύσει, ούτε καν για τις περιβαλλοντικέ παρεμβάσεις. Ε, αυτό λοιπόν περιπλέκει την κατάσταση, διότι όπω ανέφερα αυτή η εταιρεία βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι υποδικαστικά μέτρα, βασικά έχει πτωχεύσει. Ο μόνος πιθανός επενδυτής αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι το Ιταλικό κράτος. Ωστόσο ξεκίνησε διαδικασία για την ανέβρεση ιδιωτών επενδυτών. Αυτή συνεχίζεται η διαδικασία, το παρακολουθούμε με τους συνοδέλφους της DG Ανταγωνισμού και συμφωνήσαμε γιατί κάναμε και εμείς επίσκεψη επιτόπου να δούμε το ενέκταση του προβλήματος, τι μπορεί να γίνει και τι όχι. Και ε, αυτό που ε, συμφωνήθηκε είναι ότι η ρήπανση είναι το σοβαρότερο πρόβλημα. Η ρήπανση που προκλήθηκε από τη λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων την τελευταία δεκαετία πρέπει να αποκατασταθεί γιατί αυτό είναι μεγάλο βάρος για το περιβάλλον και για τον πληθυσμό που ζει εκεί. Υπάρχουν ακόμα χρήματα που μπορούν να καταβληθούν για την ώρα από το Ιταλικό κράτος ε, από τη στιγμή που οριστεί ο από το ίδιο το κράτος θα πρέπει να αναλάβει εκείνο τα, τα, τα, τα, τα, τα κόστη αυτά. 400 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσιμα. Πρόκειται για απόβλητα που βρίσκονται επί τόπου, ε, την σκόνη, τα λίματα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία και ε, όπως σας είπα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το τι γίνεται. Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για αυτές οι επενδύσεις καθαρισμού, ενώ παράλληλα, με την, ε, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίηση. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι, όπως ανέφερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως το περιβαλλοντικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνεται και αυτό στις προϋποθέσεις έγκρισης, ε, δεν έχει, δεν έχει ε, γίνει σεβαστό. Ωστόσο, αν βρεθεί ιδιώτη επενδυτή, μπορεί να αλλάξουν και τα επενδυτικά σχέδια. Και από τη στιγμή που τα επενδυτικά σχέδια αλλάξουν, τότε αυτό θα έχει αντίκτυπο και στα περιβαλλοντικά σχέδια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας ε, ελέγχουν τις προσφορές που περιλαμβάνουν και περιβαλλοντικά σχέδια. Εφόσον λοιπόν θα βρεθεί καλύτερη προσφορά, θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε το περιβαλλοντικό της σχέδιο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι οι περιβαλλοντικές ε, ρυθμίσεις να καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες και τις μελλοντικές δραστηριότητες αυτού του εργοστασίου ώστε να προστατευτεί το περιβάλλον και η υγεία του τοπικού πληθυσμού. Οι δυνατότητες της παραγωγής έχουν περιοριστεί από το 2012, πράγμα το οποίο με τη σειρά του βέβαια μείωσε τη ρήπανση. Για την ώρα λοιπόν η ρήπανση του αέρα είναι υποέλεγχο θα έλεγα Και αυτό είναι κάτι που έλαβε υπόψη η Επιτροπή. Αν όμω έπρεπε να λειτουργεί στη full το εργοστάσιο θα υπήρχαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η Επιτροπή εξακολουθεί λοιπόν να, λειτουργεί, να συνεργάζεται στενά με τις ιταλικέ Αρχές ώστε να βρει τις καλύτερες δυνατέ λύσεις για το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας είπατε τι συμβαίνει. Πολύ καλό είναι που γνωρίζουμε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά το τι συμβαίνει. Οι διαδικασίε κατά παράβαση προχωρούν. Ευχαριστούμε κύριε Λαβία μου και ε, καλή σας μέρα. Έχουμε λοιπόν τον Νικόλα Μινάση ή τον Βερμότα Φερνάρη που είναι εδώ παρόντες μπορείτε να πάρετε το λόγο σύντομα όμως γιατί πρέπει να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά σήμερα να είμαι εδώ. Πάντοτε είμαστε ε, ευτυχεί να συμμετέχουμε στη συνεδριάσεις αυτή τη Επιτροπή σα. Είναι η τέταρτη φορά που μιλάμε σε ένα χρόνο για το θέμα τη ΕΛΒΑ. Τα νέα σήμερα είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να προσθέσω μόνο ένα πράγμα γιατί όσα είπε ο πρόεδρος Λαβία και η Επιτροπή και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια πως η Ιταλία είναι ενδιαφέρουσα χώρα. Συμφωνώ μαζί σας πρόεδρε και η ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή τη φάση είναι ότι η διαδικασία πώληση των εγκαταστάσεων έχει μπλοκαριστεί και γίνεται, θα γίνει υπό τον όρο ε, της έγκρισης του περιβαλλοντικού σχεδίου του επενδυτή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εάν ο επενδυτής αγοραστής δεν υποβάλει ένα σχέδιο περιβαλλοντικό σύμμορφο προς τις ε, περιβαλλοντικές οδηγίες, δεν πρόκειται καν να εξεταστεί το αίτημα το οικονομικό, η προσφορά του οικονομική. Δηλαδή, πρώτα έρχεται το περιβάλλον και μετά η προσφορά του. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με κάθε, περίπτωση, με κάθε τρόπο την σκέψη της Επιτροπής σας στο όπως έγινε και με την ε, ε, Επιτροπή ε, που περιβάλλοντος και την αποστολή της σε εμά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ και τώρα θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. η κυρία Ευή Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που ήρθα έτσι με καθυστέρηση σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα όπου πρέπει να τρέχω ανάμεσα σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλες υποχρεώσεις και δεν άκουσα την ε, έκθεση του Προέδρου Λαβία. Απλά ε, φαντάζομαι ότι η πρόσκληση για να δοθεί σημασία τόση και φως σε αυτό την υπόθεση διαιτιολογείται από την δική μας επίσκεψη στον Τάραντα και σας ευχαριστώ για αυτή την ανακοίνωση από πλευρά τη μόνιμη αττική αντιπροσωπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την οπτική για να μπορέσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα και η Επιτροπή μα θα πρέπει να συμβάλλει και αυτή σε την επίλυση αυτού του σοβαρού θέματο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι για την επίσκεψή μας ε, στον Τάραντα και σας διαβεβαιώ ότι και η γραμματεία, αποκινούμε την γραμματεία MV, παίρνει τα στοιχεία από την ε, ε, αποστολή και τα διανέμουν σε όλους την Επιτροπή πριν πάμε εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τη την προσωπία. Και τώρα Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμόν 7. Συγκεκριμένα αναφορά 1459 Judith Klein Ουγγρική Ιθαγένειας Open Society Foundation με την υποστήριξη 12 ενώσεων σχετικά με την επένδυση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαταστάσεις για τα άτομα με αναπηρία σε ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Είναι παρούσα η αναφέρουσα. Να σας πω απλά ότι τώρα έχουμε και την αποστολή ε, στη Σλοβακία 22-23 Σεπτεμβρίου στην οποία προσβλέπουμε με υπομονησία διότι όπως γνωρίζετε αυτή η αναφορά ουσιαστικά είναι και η βάση του ενδιαφέροντος ε, που έχουμε για να επισκεφθούμε τη Σλοβακία. Κύριε Κλάιν, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στη συνάντηση αυτή ε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψής σας στη Σλοβακία. Είστε σε μια προνομική θέση γιατί η επίσκεψη και η έκθεσή σας θα δώσει σε μια ομάδα ατόμων το μεγαλύτερο δώρο, ελευθερία και αξιοπρέπεια τα θεμελιώδη δικαιώματα που τους στερήθηκαν όταν τους έβαλαν σε ιδρύματα. Αν πάτε και δείτε τα ιδρύματα και στη, συγκρίνετε τη ζωή εκεί με τη ζωή που θα ήταν δυνατή αν τους υποστήριζαν αυτούς τους ανθρώπους για να ζήσουν ανεξάρτητα μέσα στην κοινωνία, να ακούσετε τις ε, ιστορίες των, ε, πέλα, των ε, τροφίμων σε αυτά, θα δείτε τι έχουν στερήσει αυτά τα ιδρύματα από τους ανθρώπους αυτούς και μπορείτε να τους τα ξαναγυρίσετε πίσω, ασκώντας πιέσεις και εσείς προς τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις νόμιες υποχρεώσεις τους δυνάμει της σύμβασης του ΙΕ για τα άτομα με αναπηρίες. Θα δείτε λοιπόν ότι με την κατάλληλη υποστήριξη όλοι μπορούν να ζήσουν μέσα στην κοινωνία αν υπάρχει διαθέσιμη απαραίτητη υποστήριξη. Και είναι καλύτερα πάντα να ζει κανεί μέσα στην κοινωνία και όχι απομονωμένο σε ένα ίδρυμα. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τον Τραϊάν που ζει ε, σε ένα από, τα, από τους οίκους μας ε, στην ε, Κροατία. Αν έχει ήλιο εκείνη τη μέρα θα πάει να κάτσει τον ήλιο, θα βγάλει την πλούζα του. Αν βρέχει όμως θα μπει μέσα θα βγάλει το που κάψει, θα ξαναβγεί να σταθεί ε, στην ε, ε, βροχή. Είναι κοφάλαλος, τον βάλα σε ίδρυμα οι του γιατί δεν ξέρει τι να τον κάνουν, ούτε το ίδρυμα ξέρει τι να τον κάνει. Με τέτοιες δυσκολίες, ένα άτομο που δεν μπορεί να επικοινωνήσει, τι το κάνει κανείς. Αυτό που έκαναν, τι κάναν, τον έβαλαν σε απομόνωση. Για 30 χρόνια συγκεκριμένα ήταν σε απομόνωση, τον βρήκαμε εμείς, τον βγάλαμε και τώρα με όποια ευκαιρία βγαίνει έξω για να νιώσει τα στοιχεία της φύσης που ποτέ δεν μπόρεσε να τα ζήσει. Του αρέσει επίσης να πηγαίνει μακρινούς περιπάτους. Αυτά τα ανακαλύψαμε διότι ε, η επιλογή είναι η βάση για την ε, ζωή μέσα σε μια κοινότητα. Ε, να μπορεί να επιλέγει το άτομο που θα ζήσει, με ποιον, ποιοι θα είναι οι στόχοι του, τι θα φοράει, τι θα τρώει. Κάποιες φορές, σε ακραίες περιπτώσεις σαν αυτήν βέβαια, η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη ε, για την παροχή υποστήριξης, αλλά πάντοτε είναι καλύτερα ε, στην κοινωνία, μέσα στην κοινότητα και όχι μέσα σε ένα ίδρυμα. Ε, η ιδρυματική φροντίδα επιβάλλει ένα καθεστώς σε όλους. Δεν μπορεί να ρωτήσει κανεί, δεν σε ρωτάει κανεί τι θέλει, ε, ούτε για τη ζωή σου, ούτε για να φας. Δεν υπάρχουν επιλογές. Επίσης πρόσφατα συνάντησα την Ιλώνα, μια βοηθό, εργαζόταν σε ίδρυμα, τώρα όμως έχει πάρει κάποια επανεκπαίδευση για να εργάζεται σε κοινοτικά κέντρα που φιλοξενούν άτομα με αναπηρία και μου είπε ότι έχασα 20 χρόνια από τη ζωή μου εργαζόμενη σε ένα ίδρυμα. Έπρεπε να πλένω 60 άτομα τη μέρα, να τα αλλάζω. Ήταν σαν ένα, εργοστάσιο, ποτέ δεν θα ξαναπάω σε μια τέτοια δουλειά. Βλέπω τώρα ε, την ε, ανάπτυξη ε, των τρόφιμων. Βλέπω ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που ποτέ δεν φαντάζονται ότι μπορούν να κάνουν μόνοι του. Ε, μαγειρεύουν, διαλέγουν τα ρούχα που θα φορέσουν, διπλώνουν τα ρούχα τους, πηγαίνουν και επισκέπτονται φίλους, συγγενεί, έχουν χόμπι. Κάποιοι έχουν και φιλενάδα ή φίλο, έχουν δουλειέ κάποιοι, κάνουν τη δική του ζωή, είναι ευτυχισμένοι. Τώρα πράγματι αγαπώ τη ζωή μου. Το να περιορίζει κάποιος τις ελευθερίες ενός άλλου, να τον βάζει κάτω από ένα καθεστώ. είναι μια μορφή τιμωρία την κοινωνία. Αυτές τις τιμωρίες τις, θα πρέπει να τις περιορίζει στους ε, κρατούμενους, στους εγκληματίες. Πώς μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτό για άτομα με αναπηρία. Πώς θα δικαιολογήσουμε στους φορολογούμενους που χρηματοδοτούν με τα χρήματά τους. Βλέπουμε ότι αυξάνεται και ο σκεπτικισμός. Μπορούμε να δώσουμε ακόμα ένα ε, λόγο σε αυτά τα άτομα. Να τροφοδοτήσουμε τον ευρωσκεπτικισμό. Σίγουρα υπάρχουν κάποια όρια στις δικές εξουσίες, αλλά θα ήθελα να πιέσετε την Κομισιό να εγκρίνει τις συστάσεις της Ευρωπαίας Δημοσιολαβήτριας ε, που έκανε έρευνα το 2014 και συνέστησε η Κομισιόν να, συγκροτήσει ένα διαφανή προσβάσιμο μηχανισμό στο πλαίσιο του οποίου θα ερευνά η ίδια η Κομισιόν τις καταγγελίες ε, για την ε, ε, χρήση των κονδύλων κατά τρόπο που να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε βελτιώσει στου νέου κανόνε για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να μπορούν να επενδύουν χρήματα σε ιδρύματα χωρί να μπορεί να το γνωρίζει η Κομισιόν. Αν ε, μείνει ένα από αυτή την παρουσία στο μυαλό σα, θα έπρεπε να είναι το ότι 20 χρόνια που δουλεύω σε αυτό το τομέα κανένα από του πελάτε μου που έφυγε από ένα ίδρυμα δεν ζήτησε να ξαναεπιστρέψει. Ούτε ένας ας ξαναδώσουμε την αξιοπρέπεια και την ελευθερία σε αυτά τα άτομα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Thank you your Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Πραγματικά άλλαξε. Τα πράγματα καταγράφηκε ε, και πρέπει να σας πω ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται στο διαδίκτυο, άρα ξέρετε ότι ακούν και παρακολουθούν πολύ κοντά άνθρωποι από τις 28 χώρες μέλη της Ένωσης αυτά που γίνονται. Σας ευχαριστώ για την αφοσίωσή σας, για το πάθος σας, για τη συμπόνια και για την έμπνευση που μας παρέχετε. Και τώρα να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Άντορ Ούρμας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ Γιούντιτ για την εξαιρετική σου ομιλία. Θα ήθελα πολύ σύντομα να σας εξηγήσω τι έχει γίνει μετά την υποβολή της αναφοράς και να τονίσω κάποια από τα πράγματα που είπατε. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους συναδέλφους δίπλα μου από τις Γενικές Διευθυνσίες ε, Υγείας και Ρέτζιο και εκπροσωπούν μη ε, χώρες της ε, Κεντρικής Ευρώπης ε, και εγώ είμαι από την Γενική Διεύθυνση Regio αρμόδιος για θέματα τέτοιων υπηρεσιών. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα αυτό και τις δυσκολίες που συναντούν οι άνθρωποι στα ιδρύματα. Γι' αυτό τα τελευταία 5 ή 6 χρόνια έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές και στην ε, πολιτική και στους ε, κανόνες ε, των διαστροφικών ταμείων για να βρεθούν καλύτερες λύσεις για τους ανθρώπους που υποφέρουν λόγω της ιδρυματοποίησης. Πολλά από τα προβλήματα που έχουμε συναντήσει κατά τη χρηματοδότηση ιδρυμάτων στην Ανατολική Ευρώπη έχουν επανεξεταστεί. Δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα προβλήματα. Γι' αυτό, ε, κυρία Πρόεδρε, όπως αναφέρατε κατά την προπαρασκευαστική μας ε, συνάντηση, ο κανονισμός της Επιτροπής λέει σαφώς ότι δεν θα πρέπει να δαπανώνται πια πόροι στα ιδρύματα για την ανακαίνισή τους ή για νέα ιδρύματα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες εξαιρέσεις αιτιολογημένες από τα κράτη-μέλη, πρόκειται όμως πραγματικά για εξαιρέσεις. Όλα τα έγγραφα λένε σαφώς ότι δεν θα πρέπει να δίδονται χρήματα σε ιδρύματα. Η μόνη επιλογή είναι από ιδρυματοποίηση να παρέχονται υπηρεσίες στους ανθρώπους αυτούς εντός της κοινότητας. Ε, η κοινωνική φροντίδα, η υγειονομική περίθαλψη, θέσεις απασχόλησης κλπ. η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ανθρώπων με Αναπηρίες, για τα ε, δικαιώματα των ε, παιδιών. Ε, είναι σημαντικά έγγραφα αναφοράς τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών, τα οποία ουσιαστικά έχουν ενσωματωθεί στους κανόνες για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανόνες αυτούς. Εάν υπάρχει κάποια παραβίαση του νομικού πλαισίου, έχουμε κάθε δικαίωμα να ενεργήσουμε. Να διακόψουμε τις πληρωμές ή ακόμη προορατικά να σταματήσουμε την ε, διαδικασία ενός διαγωνισμού με συναδέλφους, με εμπειρογνώμονες. Ε, έχουμε συζητήσει επανειλημμένα ότι δεν θα πρέπει να ενεργεί εκ των υστέρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού, αλλά ήδη πριν να ενεργούμε προορατικά δηλαδή. Κάτι που έχει γίνει σε κάποιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπου έχει διακοπεί ο διαγωνισμός. τα μέτρα που θα στηρίζονται από τα διαφορετικά ταμεία. Συνειδητοποίησαμε ότι δεν ευθυγραμμίζονταν με τους κανόνες αυτούς και τι συμβάσει του ΟΗΕ. Μάλιστα, να σα αναφέρω ότι υπάρχει μία περίπτωση όπου ζητήθηκε να διακοπεί ο διαγωνισμός και αυτή τη στιγμή συζητιέται ακόμα το πώς μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε καλύτερα μέτρα μεταξύ άλλων και την πρόσβαση σε ε, μέτρα σε υπηρεσίες εντός κοινότητας. Όσον αφορά την απόφαση ε, του, του Ombudsman, ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της Διαμεσολαβήτριας, απαντήσαμε και είπαμε ότι ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει διαφανής τρόπος υποβολής προσφυγών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαρίστως θα παρακολουθήσουμε τις πρόσφυγες αυτές. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω. Τι γίνεται σε κάποια ιδρύματα και τι γίνεται με την έκθεση για τα διαφθορτικά ταμεία. Πάντως δεν βλέπουμε να υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην κακή μεταχείριση ανθρώπων εντός των ιδρυμάτων και ε, την ε, χρήση των διαφορετικών ταμείων. Ε, δηλαδή σε κάποια ιδρύματα ε, η κακή μεταχείριση των ε, ασθενών των έγκλειστων δεν συνδέεται άμεσα με την στήριξη από τα διαφορετικά ταμεία. Αλλά εάν δεν συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα ιδρύματα τότε θα είναι πολύ χαμηλότερο ο κίνδυνο τη κακή μεταχείρισης. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε με βάση την αρχή της αποϊδρυματοποίηση, διότι έτσι υπάρχει πολύ μικρότερος κίνδυνος ε, κακής μεταχείρισης. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι οργανώσαμε και κάποια σεμινάρια, διμερείς επαφές με κράτη-μέλη από το 2013 και μετά. Έχουμε οργανώσει σεμινάρια στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για να συζητήσουμε διάφορε πτυχές ε, των προγραμμάτων ε, των διαφορετικών ταμείων. Στην Πολωνία, στην Σεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, ε, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία έχουμε ήδη οργανώσει σεμινάρια και προβλέπονται και άλλα μέσα στους επόμενους μήνες. Πρόκειται για εξαιρετικέ ευκαιρίες να συζητηθούν οι λεπτομέρειες, το πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των προγραμμάτων του. Και αν τα κράτη-μέλη έχουν συγκεκριμένε ανάγκες και αιτήματα, πολύ ευχαρίστω τα ακούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με εμπειρογνώμονες ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομάδας ε, για την ε, αποϊδρυματοποίηση που ξεκίνησε τις εργασίες της το 2009. Έχουμε εξαιρετικές ευκαιρίες να συζητήσουμε μεθοδολογία και λεπτομέρειες της πολιτικής DI ιδρυματοποίηση ε, και της μεταφοράς ε, στην παροχή υπηρεσιών εντός της κοινότητας. Το βασικό λοιπόν εδώ είναι να αξιολογήσουμε τις ανάγκες ε, των ανθρώπων, διότι σε κάποιες περιπτώσεις συνειδητοποιήσαμε ότι η αιτιολόγηση για την επένδυση σε ιδρύματα βασίζεται σε συγκεκριμένες ανάγκες, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν σωστά οι ανάγκες. Ενθαρρύνουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν σωστά τις ανάγκες, να καταλάβουν τους ανθρώπους που έχουν τοποθετηθεί σε ιδρύματα ή που προβλέπεται να τοποθετηθούν σε ιδρύματα. Τι θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί. Αν καταλάβουμε σωστά αυτές τις ανάγκες, τότε ε, και τα διαστατικά ταμεία θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις ανάγκες αυτές. Ε, θα πρέπει να αναπτυχθεί η σχετική μεθοδολογία και κάποιες από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, κάποιοι από τους εμπειρογνωμονές μας ήδη έχουν ε, αξιολογήσει τις ανάγκες των ανθρώπων, κάτι που θα βοηθήσει στο μέλλον να επενδύουμε πιο σωστά σε υπηρεσίες ε, που να προέρχονται από την κοινότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Πρόεδρος, να δώσω το λόγο στους συναδέρφους. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Θα δώσω το λόγο λοιπόν πάλι στην κυρία Κλάιν. Α, η, κυρία Κούνεβα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δεν ήθελα να κάνω ερωτήσει, ήθελα να διαβεβαιώσω ως μέλος της αποστολής που θα επισκεφτεί τη Σλοβακία ότι συναφέροντες ότι θα είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στην επιτόπια έρευνα. Το θέμα διαχείρισης των κοντιλίων και η σπατάλη των πόρων για τα άτομα αναπηρίας είναι πολύ ευαίσθητο και θα είμαστε βέβαια ότι ε, να είναι βέβαια ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Σε ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θα πάμε ταξίδι μαζί. <laughs> Okay, now the floor goes to you, Mrs. Klein, for two minutes. Κυρία Κλάιν, έχετε ξανά το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, η ζωή σε ένα ίδρυμα παρότι μπορεί να μην κακοποιείται το άτομο, να μην ε, υφίσταται καταπεινώσει. Σίγουρα ε, συνιστά παραβίαση της ελευθερίας του των δικαιωμάτων του. Ε, στερείται τη ζωή μέσα στην κοινωνία. Ένα αυτό. Και δεύτερον, το έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι υπάρχει ένας κίνδυνος. Τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη τέλος πάντων, να μιλήσουν για αποϊδρυματοποίηση βάζοντας αυτόν τον τίτλο σε κάποια προγράμματα που δεν ε, αφορούν ουσιαστικά την αποϊδρυματοποίηση αλλά τη δημιουργία μικρότερης κλίμακας ιδρυμάτων. Δεν είναι αυτό η αποϊδρυματοποίηση όμως, απλά το να τους βάλουμε σε ένα μικρότερο χώρο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. I thank you very much. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και πράγματι το έχουμε αντιληφθεί αυτό χθε, το είπε και ο κύριο Σούρμο. Ήμασταν σε μια προπαρασκευαστική συνάντηση και με την κυρία Γκέρλεν που είναι η προϊσταμένη του τμήματο για τη γάμα δέλτα, την αρμόδια της Κομισιόν και πραγματικά Είδαμε την αποφασιστικότητα, παρακολουθείτε στενά το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στη διάρκεια αυτής της διερευνητικής επίσκεψης ώστε να μην παραβιάζεται πλέον η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους να μην επικρατήσει στέση ελευθερία του. Σα ε, εγγυώμαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στη διάρκεια αυτή τη επίσκεψη και σα ευχαριστούμε θερμά για την αφοσίωσή σα, ε, την προσήλωσή σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Και πάλι σα ευχαριστώ και που ήρθατε εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι με έχει συναρπάσει αυτή η επίσκεψη και ξεχνάω τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, ουσιαστικά η αναφορά που είναι και η βάση αυτή την επίσκεψη παραμένει ανοιχτή. Θα αναφέρουμε στους υπόλοιπους συναδέλφους ε, της Επιτροπής μας και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλους ε, για τα πορίσματα αυτής της επίσκεψης. Άμα τη επιστροφή μας. Επίσης έχει πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι εδώ για να εξασφαλίσει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό παρακολούθησης της χρήσης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και όπως είπατε και εσείς, το θέμα είναι η πραγματική αποϊδρυματοποίηση, όχι η δημιουργία μικρότερων ιδρυμάτων, αλλά να ξαναδώσουμε πίσω την ελευθερία τους σε αυτά τα άτομα. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό θα δούμε και εμείς σε βάθος. Μέχρι τότε παραμένει βέβαια ανοιχτή η αναφορά. Σας ευχαριστώ και πηγαίνω στο σημείο 8 της μερίσιας διάταξης. Είναι η αναφορά 0509 και η 169 μαζί. Είναι οι αναφέροντες παρόντες, αλλά θα δώσω καταρχάς λοιπόν το λόγο στη Σίλβια Μακοβίακ και στον Αντάμ Σπρεσίνσκι και οι δύο λοιπόν έχετε το λόγο αλλά το πολύ για πέντε λεπτά. That is in total, so try... Συνολικά πέντε λεπτά. Μοιραστείτε τον αυτό το χρόνο. Dzień dobry, nazywam się Sylwia Maćkowiak. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε στη σημερινή συνεδρίαση. Ε, έχουμε την Ένωση Σάλνταμ που που ε, συγκεντρώνει τους κατοίκους ε, αρκετών δήμων της Νότιας Πολωνίας. Έχουμε συγκεντρώσει λοιπόν υπογραφές κατά της κατασκευής ενός ε, ορυχή ανοιχτή εξόριξης λιγνίτη στην περιοχή μας. Ε, οι κάτοικοι, οι γεωργοί, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταποίηση ζωικών προϊόντων απειλούνται. Οι επενδυτές θέλουν να, να καταστρέψουν 10.000 εκτάρια κατασκευάζοντας αυτό το ορυχείο ανοιχτή εξόρυξης. Τα σπίτια μας, τα αγροκτήματά μας, τα εργοστάσια μας, οι δουλειές μας θα εξαφανιστούν και θα είναι κάτι που, που μετά θα τελειώσει επιστρεπτεί. Υπάρχουν περισσότερες ε, θέσεις απασχόλησης που θα καταργηθούν μετά από την κατασκευή αυτού του ορυχείου λιγνίτη από ό,τι θα δημιουργηθούν. Οι αρχικές εργασίες διερεύνησης ξεκίνησαν τις 11 Μαΐου του 2011 όταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος έδωσε την άδεια στην ε, εταιρεία ΠΑΚ για να προβεί στις πρώτες ε, ε, εργασίες αναγνώρισης στις περιοχές του Άπονιας και Σκοβίτσε. Η απόφαση αυτή λήφθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας και της ιδιοκτησίας. Από τις αρχές διαμαρτυρόμεθα κατά αυτής της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος. Διότι οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Θα κατασκευαστεί αυτό το ορυχείο Έχουμε διαμαρτυρηθεί ενώπιον των δημόσιων αρχών, ενώπιον των δικαστηρίων, έχουμε ε, διαμαρτυρηθεί και στους δρόμους. Έχουν υπάρξει σφάλματα διαδικασίες τα οποία ποτέ δεν διορθώθηκαν. Οι αρχικές ε, γεωτρήσεις ξεκίνησαν κατά, ε, μάλλον ενάντια στη γνώμη των ιδιοκτητών των ε, ε, γεών. Ε, το 2015 αυτό το έγγραφο που βασίζεται στα σφάλματα διαδικασίας είναι αυτό που εγκρίθηκε από τον Υπουργό, πράγμα που οδηγεί στο ότι αυτά τα κοιτάσματα λεκνίτη είναι πλέον προστατευόμενα. Ε, μέχρι τα τέλη αυτού του έτους ε, τα αποθέματα λιγνίτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της ε, χωροταξίας στην περιφέρειά μας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα επενδύσεων ή συναλλαγών σε ακίνητες περιουσίες στην περιφέρειά μας, γιατί φυσιμένει αυτό καταδίκη σε θάνατο. Ποιος θέλει να δεσμεύσει τα χρήματά του όταν ξέρουμε ότι σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει πλέον ψυχή σε αυτή την περιφέρεια και θέλουμε να δράσουμε τώρα για να ε, τηρηθούν και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα της του Ευρωπαϊκού Χάρτη. Το άρθρο 7 ήδη έχει παραβιαστεί στο χάρτη αυτό. Σήμερα ζούμε μέσα στην αβεβαιότητα όσον αφορά τη μοίρα μας και το μέλλον μας. Δεν ξέρουμε τι θα μας περιμένει στο μέλλον ποιο θα είναι το μέλλον μας σε 5-10 χρόνια. Στο άρθρο 17 επίσης έχει παραβιαστεί διότι οι γεωτρήσεις έχουν γίνει ενάντια στην άποψη των ιδιοκτητών των ε, γεών επί των οποίων έγιναν οι γεωτρήσεις. Υπάρχουν δικαστικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει αλλά ε, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και επίσης η απόφαση έχει ήδη ληφθεί το 2014 όσον αφορά την προστασία αυτών των επαθεμάτων λιγνίτη. Παρά το ότι έτρεχε διαδικασία δικαστική, παρά την παραβίαση αυτών των διαφόρων αρθρων, εάν προστατευτούν αυτά τα αποθέματα λιγνίτη σήμερα, σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε και στην επόμενη φάση της κατασκευής του ορυχείου. Και γι' αυτό και κάνω έκκληση σε όλους τους βουλευτές σήμερα. Πρέπει τώρα να δράσουμε. Θα είναι αργά όταν θα, ξεκινήσουν, θα ξεκινήσει η εξόριξη και όταν ε, χιλιάδες άνθρωποι θα χάσουν τα σπίτια τους στο περιβάλλον δε θα ε, επιβαρυνθεί αναπότρεπτα. Θα είναι μια τεράστια απώλεια. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς θα ήθελα να σας ε, συστηθώ. Λέγομαι Άντα Μαζένσκι και είμαι ένας εκπρόσωπος των τοπικών αρχών. Δεν αντιπροσωπεύω όμως μόνο μία τοπική αρχή, αλλά όλους τους Δήμους που απειλούνται από αυτό το ορυχείο. Και θα ήθελα σήμερα να ε, υπογραμμίσω την αβεβαιότητά μου, την αβεβαιότητά μου η οποία, για, για την ε, ε, βαραίνει όλους τους ανθρώπους της περιοχής. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μια διαδικασία που δεν είναι καν ολοκληρωμένη. Όλες οι γεωτρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ε, 167 από τις 381 που έπρεπε να γίνουν. Ε, λήφθη μια απόφαση το 2015 επί τη βάση πληροφοριών και πολλοί εμπειρογνώμονε το υπογραμμίζουν αυτό. Η Επιτροπή που, ασχολείται με τα υδρολογικά ζητήματα θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί και αυτή με αυτό το θέμα και δεν ζητήθηκε η γνωμοδότησή της. Το 2015 ο Υπουργό ακύρωσε όλη τη διαδικασία διαδικασία σε σχέση με τη δική μας διαμαρτυρία. Εμείς σήμερα σας ζητάμε βοήθεια γιατί βασιζόμενοι στην νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον, όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, θα πρέπει πραγματικά να σεβαστούμε το τοπικό δικαίωμα των ε, δήμων ε, της περιοχής, ε, πράγμα που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το κράτος αναμειγνύεται στις δικές μας αρμοδιότητες και δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία που προχώρα ενάντια στην γνώμη μας. το Γεωλογικό Ινστιτούτο το κρατικό έχει ήδη δημοσιεύσει ένα έργο στο οποίο ε, λέει ότι αυτά τα αποθέματα ήδη έχουν αναγνωριστεί. Προχωράει η διαδικασία δηλαδή από εκείνη την πλευρά και κατά τη γνώμη μας αυτό δεν συμφωνεί με το άρθρο 4.6 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις ε, τοπικές ε, κοινότητες θα έπρεπε να έχει γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες όταν λαμβάνεται μια αναπόφαση η οποία άμεσα επηρεάζει την ζωή του, των πολιτών. Αυτή η διαδικασία έπρεπε να έχει σταματήσει. Ήδη σήμερα έχουμε απόλυος. Ε, ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά καταστροφή για τους Δήμους μας. Ευχαριστώ λοιπόν την ε, Επιτροπή που έστειλε την επιστολή στις πολωνικές αρχές. Δυστυχώς η αντίδραση ήταν εξαιρετικά αρνητική από ό,τι μπόρεσα να καταλάβω και ελπίζω πως σήμερα θα ασχοληθείτε και πάλι με αυτό το θέμα ε, και φυσικά σας καλώ να έρθετε στην περιοχή μας γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να σας αποδείξω επί τόπου πώς έχουν τα πράγματα και να σας δείξω τι συμβαίνει. Ε, θα ήθελα ε, να διαρτηρηθεί λοιπόν ανοιχτή αυτή η αναφορά ώστε να αποφύγουμε ε, την καταστροφή του, της κληρονομιάς μας λόγω αυτής της απόφασης. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε και στον Τόμας Πάβελ Αρμπεύσκη που είναι εδώ για την αναφορά 169. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Οι συνάδελφοί σας μίλησαν λίγο πολύ. Ε, ε, παρακαλώ λοιπόν εσείς να είστε πιο σύντομος. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ θα σας παρουσιάσω τη θέση της δικής μας ε, οργάνωσης που είναι η εταιρική σκέψη για την οικολογία, υπέρ της οικολογίας. Στηρίζουμε τους προλαλήσαντες και τις προσπάθειές τους προσπαθούμε να συνεργαστούμε με την Ένωση που έχουν δημιουργήσει αλλά και με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας μας. Δεν μπορούσαν να είναι όλοι παρόντες στις Βρυξέλλες βέβαια, αλλά εξ ονόματος όλων των μελών της οργάνωσής μας θέλω να πω ότι είμαστε κατά αυτού του σχεδίου κατασκευής λιγνητορυχείου θα είναι τραγική μια τέτοια εξέλιξη και για τους γεωργούς, ε, γιατί η εκμετάλλευση σμάτων λιγνίτη θα έχει ως αποτέλεσμα την συμπίεση του υδροφόρου ορίζοντα και η υποβάθμιση του εδάφους. Ε, δεν θα μπορούν δηλαδή οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι επιχειρήσεις πλέον ε, να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους και μιλούμε για χιλιάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σήμερα η παρουσία των κοιτασμάτων ήδη είναι ε, αντική διότι είναι υποπροστασία, έχουν σταματήσει επενδύσεις, γι' αυτό και αυτή η περιοχή της Ευρωτής Πολωνίας, ε, όπως λέγεται, έχει υποφέρει ε, από οικονομικής πλευράς. Εμείς έχουμε συμπεριλάβει όλα τα επιχειρήματα στην αναφορά μας, την 169 από το 2015 και ελπίζω να μπορέσετε να την δείτε ευνοϊκά. Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Πρώτος, ευχαριστώ όλες και όλους που μας μεταφέρατε τις εμπειρίες από την πραγματικότητα που ζείτε και τις πεπιθήσεις σας και τα συναισθήματά σας. Στρέφομαι στην Άννα Στεγιασκόφσκα ή κάπως έτσι από την Κομισιόν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και τους ε, αναφέροντες θέλω να ευχαριστήσω και θέλω να υπογραμμίσω ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τον Μάρτιο του 2015 που σημαίνει ότι προς το παρόν η μόνη δράση που έχει αναλυφθεί είναι οι γεωλογικές μελέτες ε, για τα κοιτάσματα λιγνίτη. Μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε να υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο για το περιβάλλον, άρα η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απαιτεί την ανάληψη δράση. Βέβαια, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτή τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου, προτού δοθεί άδεια για να ξεκινήσει αυτή η επένδυση, τα άτομα που θέλουν να φτιάξουν αυτό το λιγνητορυχείο θα πρέπει να υποβάλουν μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Οι επενδυτές υποχρεούνται δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπεται να δημοσιοποιήσουν, να δημοσιεύσουν αυτή τη μελέτη. Εμείς θα αναλύσουμε όλους τους πιθανούς αντικτύπους Μια ε, μιας τέτοιας επένδυσης στο περιβάλλον. Έχουμε και το Natura 2000 γιατί υπάρχουν περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000 και οι οποίες πλήττονται από αυτή την επένδυση. Όλα αυτά τα στοιχεία θα τα λάβουμε υπόψη προτού λάβουμε την τελική μας απόφαση. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και ο εντόπιος πληθυσμός θα δώσει τις απόψεις, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να υποβάλουν παρατηρήσεις. Και αυτές οι παρατηρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι η οδηγία για τις μελέτες αντικτύπου περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε εθνικό επίπεδο. Η πολωνική κυβέρνηση θέλει να συνεργαστεί με τις ε, ΜΚΟ. Και αυτόματα, θα έλεγα σχεδόν, οι ΜΚΟ μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Στην ε, περίπτωση αυτή λοιπόν και σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες και δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η Ποιο θα είναι ο αντίκτυπο αυτή τη επένδυση στο περιβάλλον, δεν ξέρουμε ακριβώ τι προβλέπει ο επενδυτή. Είναι λίγο ακόμα ασαφή τα πράγματα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο σε συναδέρφους που άκουσαν προσεκτικά όλα όσα υπόθηκαν. Ε, κύριε Πτέρα, πρώτη στον κατάλογο των ομιλητών. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, εδώ πρόκειται για μια περιοχή γεωργική όπου η γεωργία ασκείται με πολύ σύγχρονο τρόπο, με πολύ ανεπτυγμένη δραστηριότητα. Εδώ και χρόνια η γεωργική παραγωγή είναι πολύ ανεπτυγμένη ε, και η βιομηχανία τροφίμων έχει έντονη παρουσία στην περιοχή αυτή. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, της πολωνικής οικονομίας και μάλιστα πολλά ανέκδοτα ε, στην ε, χώρα μου κάνουν λόγο για τους ανθρώπους αυτής της ε, περιοχής, Greater Poland, Μεγάλης Πολωνίας, πόσο οικονόμοι είναι, πόσο καλά ξέρουν να διαχειρίζονται τα οικονομικά κτλ. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε αυτήν την νέα επένδυση για ένα υπαίθρο λιγνητορυχείο. Πολύ ξεκάθαροι αναφέροντες και σημείο προς σημείο μας εξήγησαν τις επιπτώσεις που θα είχε η κατασκευή αυτού του λιγνητορυχείου μας μίλησαν και για τα διάφορα διαδικαστικά προβλήματα που ανέκυψαν και γι' αυτό θα πρέπει να απευθυνθούμε στην πολωνική κυβέρνηση ζητώντας να δώσει πληροφορίες σε σχέση με όλα τα προβλήματα που ανέκυψαν μέχρι στιγμής. Όλα τα διαδικαστικά ασφάλματα, ελλείψεις και όλα τα άλλα στοιχεία. Φαντάζομαι ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να συντάξουμε αυτή την επιστολή γιατί έχουμε όλες τις πληροφορίες από τους αναφέροντες και στην επιστολή μας μπορούμε να ζητούμε πληροφορίες για, για τη φάση ανάπτυξης του σχεδίου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και αν μέχρι στιγμής έχουν τηρηθεί οι ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Πολεμικού Δικαίου. Ζητώ λοιπόν να παραμείνει ανοιχτό το θέμα. Είναι ανοιχτό το ζήτημα, δεν μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν την αναφορά. Ευχαριστώ. η Μαγκρέτε, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ σήμερα. Έχουμε δει και σε άλλες συνεδριάσεις ε, τα ωραία μέρη της Πολωνίας και πόσο ευχαριστημένοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να διασώσουν αυτές τις ε, ωραίες περιοχές. Είναι εξωφρενικό αυτό που βλέπουμε εδώ. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην φτάσουμε στην εκροψία, να πεθάνουν όλοι και εμείς απλά να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Και δεν ε, γνωρίζουμε ακόμα αν πρόκειται για παραβίαση των κανόνων ε, των περιοχών Natura 2000. Αυτό θα πρέπει να διαπιστωθεί αλλά δεν έχει ληφθεί καθόλου η ε, οδηγία για τις ε, περιβαλλοντικές μελέτες επιπτώσεων. Και ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι σαν να ακούω την ε, κυβέρνηση της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Και ακόμα και αν δεν έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει διαδικασία σε επιπαραβάση, επειδή δεν έχουμε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, όταν μιλάμε για τις ε, περιοχές Natura 2000 ε, και τις ε, εκθέσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, είναι ότι είναι σαφές ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. και οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ θέλουν να σώσουν το μέλλον της Πολωνίας. Και στην Ανατολική η Γερμανία είδα τι κάνουν τα υπαίθρια ορυχεία. Το πώς καταστρέφεται το περιβάλλον ε, και πόσο επιβλαβές είναι για τους κατοίκους. Ε, Λοιπόν, ε, είναι πολύ θετικό που θέλετε να προστατεύσετε τη χώρα σας ε, και να αποφύγετε τους κινδύνους από αυτήν την πολύ βραχυπρόθεσμη, ε, μάλλον την οικονομία που δεν κοιτάει μακριά. Φυσικά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Przepraszam za spóźnienie, ale mam dwie Ναι, κοιτάξτε. Υπάρχουν ένα σωρό επιτροπές που συνεδριάζουν ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο να είμαστε πανταχού παρόντες. Τώρα, συμφωνώ με την Ιουλία ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, να στραφούμε στο Πολωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και να ζητήσουμε περισσότερες εξηγήσεις. Δυστυχώς στην Πολωνία λέμε συχνά ότι οι Πολωνοί ε, βάζουν μυαλό μόνο κατόπιν εορτής. Ε, όμως ε, εδώ πρέπει να βιαστούμε, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι συνέπειες ε, λειτουργίας ενός τέτοιου ρηχείου. Δεν είναι μόνο τα 25 εκτάρια, αλλά πρόκειται για τον αντίκτυπο σε μια ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Σίγουρα ο αντίκτυπος ε, σε αυτή τη τόσο γόνιμη γη θα είναι πολύ αρνητικός. Ε, δεν θέλω να επεκταθώ πολύ, αλλά θέλω πραγματικά να στηρίξω την ε, αναφορά αυτή. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αποφύγει το θέμα, αν και από νομική πλευρά δεν έχει πάτημα για να το κάνει αυτό. Όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι εδώ Ευρωπαίοι πολίτε. Και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο εμεί είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του πληθυσμού και να παίξουμε το ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στις ενώσεις των πολιτών ε, και την πολωνική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καθότι ήθελα να πω πολλά από αυτά που ήδη υπόθηκαν καλύπτηκα, αλλά θα ήθελα επίσης να σας ε, θυμίσω την αναφορά για την περιοχή Ροζάλια ανάμεσα στην ε, χώρα μας ε, και την Γερμανία και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές ε, από τα υπαίθρια λινητορυχία. Συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Πτέρα να στείλουμε επιστολή. Είχαμε μια διερευνητική επίσκεψη που είχε να κάνει με τα ποτάμια στην ε, Ισπανία Εάν δούμε και εδώ παρόμοιες ε, συνέπειες, αυτό θα αποτελέσει καταστροφή και στην Ανατολική Ευρώπη. Ούτε καν να σας μιλήσω για την Ισπανία. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τυρίψ. Ε, Πώς προφέρετε το όνομά σας. Ξύπ. Δεν θα το επαναλάβω. Τα δύο γράμματα το ρο και το ζω ε, ε, προφέρονται ζ. Όπως και να έχει ωραίο όνομα, σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πιο εύκολο να λέτε με το άλλο όνομα, Ένζο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έρχομαι από αυτή την περιοχή. Ξέρω πάρα πολύ καλά το μέρος. Ξέρω πάρα πολύ καλά που προγραμματίζεται να η κατασκευή αυτού του ορυχείου λιγνίτη. Πρόκειται για μια περιοχή με πολύ μακρά παράδοση. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι μια περιφέρεια για την οποία γνωρίζουμε εδώ και 100 χρόνια τουλάχιστον ότι κρύβει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιγνίτη ε, κανείς μέχρι στιγμής δεν τόλμησε να αρχίσει να εκμεταλλεύεται αυτά τα κοιτάσματα στην ε, λόγω περιοχή. Γι' αυτό και με εκπλήσει αυτή η απόφαση που έχει ληφθεί τώρα. Αυτό σημαίνει την καταστροφή των καλύτερων γεωργικών γεών και ολόκληρης ε, της ε, περιοχής ε, της ευρύτερης Πολωνίας του, του Νότου. Θα καταστραφεί όλη η περιφέρεια. Επίσης θα πρέπει να πω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση όχι μόνο από πλευράς ε, των ε, ε, πολιτών αλλά και από τους τοπικούς συλλόγους και ενώσει. Ίσως να ήταν δύσκολο γιατί, να το καταλάβετε γιατί εδώ έχουμε μόνο εκπροσώπους ενός από, τα δύο, τους δύο νομούς. Όμως όλες οι τοπικές και περιφερειακές ενώσεις και συνεταιρισμοί είναι αντίθετοι με αυτό το project. Μάλιστα, ε, έχουμε μία, ένα ψήφισμα από όλους τους τοπικούς ηθήνοντες ότι απορρίπτουν την εκμετάλλευση του κοιτάσματος αλλά και την δυνατότητα κατασκευής αυτού του ορυχείου. Ακούσαμε όμως και ένα άλλο επιχείρημα μέσα στην αίθουσα. Σήμερα υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις τοπικές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην περιοχή. Δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρω τα ονόματά τους ούτε να τους κάνω διαφήμιση. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτοί, αυτά τα μεγάλα, οι μεγάλες εταιρείες ε, ε, παίρνουν αποφάσεις να μην επενδύσουν άλλο ή να αποσύρουν τις επενδύσεις τους σε περιφέρεια αυτή, ενώ θα ήταν πολύ ωφέλιμα επενδύσεις από οικονομική λόγω αυτού του project. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να συμφωνήσουμε με την πρόταση της κυρίας Πιτέρα και ο αυτή η αναφορά να μείνει ανοιχτή και ότι θα πρέπει να ε, γράψουμε στην κυβέρνηση ώστε να απαντήσει σε σχέση με όλα αυτά τα επιχειρήματα που παρουσίασαν οι δύο ενώσει που είναι σήμερα εδώ. Ναι, σημειώνω το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύεται εδώ αυτή τη στιγμή. Και τώρα επιστρέφω στους αναφέροντες. Ένας από σας αποφασίστε μεταξύ σας ποιος από όλους, θα συνοψίσει σε δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, για να δούμε ποιος θα πάρει το λόγο τώρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα, αλλά να... δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα εγώ να μιλήσω για όλου, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μα όμω αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχουν εγκριθεί κάποια έγγραφα παρά τι διαμαρτυρίε μα. Ε, και σήμερα η έγκριση αυτών των εγγράφων μας φέρνει στην εξής κατάσταση. Ε, αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις τοπικές αρχές Όσον αφορά την χωροταξία θα πρέπει να συμμορφωθούν. Δηλαδή σήμερα δεν μπορούμε πλέον να, να χτίσουμε οτιδήποτε ε, σε αυτές ε, τις γέες. Ε, για 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα δεν μπορεί να κατασκευαστεί τίποτα, κανένα κτίσμα. Ήδη αυτό έχει ξεκινήσει λοιπόν. Η καταστροφή αυτή έχει ξεκινήσει. Και να κάνω άλλη μια έκκληση από πλευρά Ναι, η περιβαλλοντική πτυχή είναι πολύ πιο σημαντική εδώ, αλλά δεν είναι η μόνη. Σήμερα θα πρέπει να έχουμε μια ευρύτερη εικόνα και να λάβουμε υπόψη όλες τις αρνητικές πτυχές αυτής της κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να προσπαθήσω να συνοψίσω. Θα αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά αυτή, διότι συνεχίζεται το πρόβλημα. Θα στείλουμε επιστολή στην ε, κυβέρνηση της Πολωνίας, όπου θα αναφέρουμε ιδιαίτερα ότι θα πρέπει να μας απαντήσει σωστά ο Υπουργός ε, Περιβάλλοντος. Ε, θα πρέπει να μας δώσει πληροφορίες σχετικά με το αν υπήρξε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ε, και εάν ναι, ποια είναι τα συμπεράσματα, εάν όχι, γιατί όχι. Επίσης, να εκφράσουμε το φόβο μας ότι θα έχουμε υπερβολική ε, εκμετάλλευση της φύσης στην περιοχή αυτή που είναι γεωργική περιοχή. Πιστεύουμε ότι θα καταστραφεί η γη. Επίσης πιστεύουμε ότι είναι κοντόφθαλμη η ε, πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και να τονίσουμε ότι περιμένουμε σύντομα απάντηση. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στις Βρυξέλλες. Ελπίζω ότι θα περάσετε ένα ωραίο απόγευμα στις Βρυξέλλες και αγοράστε σοκολάτα. Η σοκολάτα των Βρυξελών είναι καλύτερη από τις ε, Πολωνίες. Σας εύχομαι να περάσετε καλά και θα είμαστε σε επαφή πάνω στο θέμα αυτό. Προχωρώ τώρα στο επόμενο θέμα, το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. Αναφορά 1160 του 2009, αναφορά 1246 του 2010 και αναφορά 1501 του 2010. που έχει να κάνει με την ε, παραβίαση κοινωτικής νομοθεσίας ε, κατά την ε, κατάσταση αιωλικών πάρκων στην μεθοριακή περιοχή της Τσεχίας. Η αναφέροντες δεν είναι παρόντες. Ελπίζω να παρακολουθούν τη συζήτησή μας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να επαναλάβω τις βασικές πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα και το τι έχει κάνει η Επιτροπή μέχρι τώρα. Πρόκειται για ένα έργο κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. Έχουμε 18 ε, ανεμογεννήτριες 3 ε, ε, ΜΒ και συνάδει με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης εφαρμόζεται η σύμβαση ΕΣΠΟ διότι ε, έχει διασυνορικές επιπτώσεις ε, και επίσης ε, υπόκειται στο άρθρο 6.3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η έγκριση ξεκίνησε το 2009 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αναμένεται όμως να ολοκληρωθεί φέτος. 19 Απριλίου του 2013 ολοκληρώθηκε η, με, ε, μελέτη η έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τη ζεχική νομοθεσία και το συμπέρασμα ήταν ότι θα έχει ε, περιορισμένες συνέπειες στο περιβάλλον. Οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν τον Ιούλιο 2010 για την κατασκευή του έργου και Οι Γερμανοί πολίτες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δημόσια διαβούλευση που οργανώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου του 2013 στην Τσεχία. Από τους 30 συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση περίπου οι 15 ήταν Γερμανοί. Ήδη το 2013 ολοκληρώθηκαν ε, οι εκτιμήσεις και για το Natura 2000 ε, και σκοπός είναι να υπάρχει ευρωπαϊκή συνένεση και αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που δεν βασίζεται στο δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρόκειται για διαδικασία παρέκκλησης από το τσεχικό δίκαιο που θα ολοκληρωθεί φέτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο συμμορφώνεται το έργο με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ήδη ενημερώσει πέντε φορές την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις εξελίξεις σε σχέση με το έργο αυτό. Δεν ε, υπάρχει όμως καμία ένδειξη ότι θα εγκριθεί ε, παραβιάζοντας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το έργο αυτό. Ευχαριστώ. Ε, δίνω το λόγο στους συναδέλφους. Μάρκαρετε, παρακαλώ. Ένα γενικό σχόλιο. Νομίζω ότι καλό είναι όλοι να το έχουμε υπόψη σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση, την προηγούμενη αναφορά για παράδειγμα. Ότι δηλαδή ακόμη και μια τεράστια ανεμογεννήτρια αν αποφασίσεις ότι δεν τη χρειάζεσαι μπορείς να την αφαιρέσεις, να την απομακρύνεις και η φύση ε, ξαναβρίσκει την προηγούμενη μορφή της. Δεν δημιουργεί δηλαδή ζημιά ε, στο περιβάλλον η ανεμογεννήτρια. Βέβαια, οι πολύ μεγάλες ανεμογεννήτριες ε, κινούνται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς. Το έχω δει στη Δανία. Δεν επηρεάζουν τόσο το τοπίο όσο οι πιο μικρές. Άρα είναι πιο εύκολο και για τα πουλιά. Και είναι και πολύ ψηλά και δεν τις βλέπεις. Τώρα ελπίζω να γίνει σωστά η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Πού θα τοποθετηθούν επίσης είναι σημαντικό. Δηλαδή μπορείς να αποφύγεις διαδρομές που παίρνουν τα πουλιά. Έχω δει κάποια σχέδια στη Βουλγαρία για παράδειγμα. Βέβαια, Υπάρχει και η άλλη τάση να κάνει κανεί επιλογή την καλύτερη δυνατή θέση. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να πάρει στη δεύτερη, τρίτη καλύτερη επιλογή. Πρέπει να τα λάβετε και αυτά υπόψη, γιατί κάποιε φορέ ε, δεν λαμβάνεται αυτό υπόψη. Γίνεται η μελέτη αντικτύπου. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να γίνει πιο κομψά το έργο και επιλογή. Καλό είναι να γίνει και μια μελέτη περιφερειακού αντικτύπου, όχι μόνο εθνική. Από ό,τι έχω μάθει όμως, έκαναν και οι Γερμανοί αξιολόγηση, μας συμμετείχαν σε αυτή την αξιολόγηση. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε τόσο πολύ αυτό το project, ε, γιατί δεν είναι για την αιωνιότητα και είναι και καλό για το περιβάλλον και το κλίμα κτλ. Κύριος Μπέκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι και εκπρόσωποι της Κομισιόν, πολύ σύντομα θα ήθελα με λίγο χιούμορ να διατύπωσω τη θέση μας. Ε, δεν λυπάμαι ούτε την Κομισιόν ούτε εμάς που πέμπτη φορά ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, διότι πρόκειται για δική μας ευθύνη να παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή και εκτιμώ και τη δουλειά της Κομισιόν στο θέμα αυτό. Έχοντας ε, ακούσει αυτά που ακούσαμε, μόνο ένα ε, ξεκάθαρο συμπέρασμα υπάρχει, να παραμείνει ανοιχτή και περιμένουμε ε, την επόμενη συνάντηση εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πίτερ. Δεν ζήτησε το λόγο, νόμιζα ότι τον ζήτησε. Ελεονόρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ παίρνω το λόγο μόνο για να επαναλάβω την ανάγκη να γίνει σωστά η μετάβαση προς τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, αυτό είναι ανάγκη όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, χωρίς όμως να αποκλίνουμε από τις οδηγίες που προστατεύουν το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα την οδηγία περί habitat και πτηνών. Όπως είπε σωστά και η συνάδελφος να είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η ε, αναφορά ώστε να φροντίσουμε ότι οι οδηγίες εφαρμόζονται σωστά χωρίς καμιά εξαίρεση και παρέκκληση. Και επιπλέον, εάν υπάρχουν ακόμα ε, διαδικασίες που είναι υπό εξέλιξη, ακόμα παραπάνω αυτή η έκθεση θα πρέπει να μένει ε, ανοιχτή. Εμείς ε, πόσο κατανοούμε και στρέφουμε στην Κομισιόν, δεν γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα τρέχει ακόμα το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Και αν θέλουμε να το διατηρήσουμε ανοιχτό μέχρι ότου να έχει ολοκληρωθεί το πιλωτικό πρόγραμμα και αξιολογηθεί και μετά να δούμε τι έγινε, να κάνουμε αξιολόγηση. Μπορείτε αυτό να μου το αποσαφηνίσετε. Πόσο καιρό προτίθεστε να διατηρήσετε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, ναι. Η παράβαση μπορεί να εντοπιστεί μέχρι ότου αδειοδοτηθεί το project. Η Κομισιόν απλώς παρακολουθεί για την ώρα μέσω πιλωτικού προγράμματος. Η διαδικασία αδειοδότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Οπότε φέτος θα πρέπει η Κομισιόν να αποφασίσει είτε ότι το πρόγραμμα θα σταματήσει είτε ότι θα ανοίξει η διαδικασία κατά παράβαση. Η Κομισιόν είναι της άποψης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει παράβαση. Μάλιστα. είτε θα συνεχιστεί το πιλωτικό πρόγραμμα, είτε θα ανοίξει η δικασία κατά παράβαση. Έτσι θα το κρατήσουμε ανοιχτό μέχρι ότου να γνωρίζουμε και εμείς θα είμαστε σε επαφή με την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε. Can we move to the next item, which is number 16 on the agenda? Πάμε στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης είναι η 1555 του 2012, ο αναφέρον δεν είναι παρόν. Και γι' αυτό και στρέφομαι άμεσα στην Κομισιόν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τονίσω τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό το project και το προηγούμενο. Εδώ αυτό το project είναι ήδη κατασκευασμένο στην Δυτική στο δυτικό σύνορο της ε, Τσεχίας, στα σύνορα με την ε, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, είναι πιο μικρό αυτό το πρόγραμμα. Είναι πέντε ε, ανεμογεννήτριες σε 2 μεγαβάτ έκαστη ε, και αυτό έχει γίνει αξιολόγηση σύμφωνα με το Natura 2000 η οποία όμως σταμάτησε στην φάση του screening οπότε και αποφασίστηκε ότι το project αυτό δεν θα είχε αντίκτυπο διασυνοριακό ε, και ότι δεν θα είχε ε, επιπτώσεις Natura 2000. Γι' αυτό και ολοκληρώθηκε η ιδιοδότηση το 2013 και προχώρησε έχει διγίνει, Η Κομισιόν έλεγξε την αναφορά, οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για το θόρυβο, τα επίπεδα θορύβου, στην τεκμηρίωση που έχουμε στη διάθεσή μας ε, ε, στο τσεχικό site που ενημερώνει για αυτό το project υπάρχει μια μελέτη για το θόρυβο που λέει ότι τα γερμανικά στάνταρ για το θόρυβο δεν έχουν παραβιαστεί, ούτε και τα τσεχικά στάνταρ για το θόρυβο από την άλλη πλευρά. Ε, Επίτα λέει ότι έχει επιπτώσεις στον τουρισμό και τα επιπτώσεις ε, στον τουρισμό δεν έχουν καμία σχέση με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για μας δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ότι έχει υπάρξει παράβαση της νομοθεσίας Natura 2000 και το project σωστά αδειοδοτήθηκε. Σας ε, ευχαριστώ. Πίτερ. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρατήρηση και μετά ε, να κάνω μια που αφορά συγκεκριμένη να, αυτή την υπόθεση. Να ευχαριστήσω τους ε, αναφέροντες και όσον αφορά ε, διασυνοριακές υποθέσεις υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας Στην προηγούμενη υπόθεση είδαμε ότι από νομικής πλευράς έγιναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν, αλλά ε, πρέπει να δούμε, έχουν γίνει οι σωστές προσκλήσεις, ε, υπάρχουν τα έγγραφα στην γλώσσα που πρέπει. Ήδη στο προηγούμενο έργο είδαμε ότι υπάρχει έλλειμμα επικοινωνίας ε, και οι πολίτες και από τις δύο πλευρές των συνόρων ε, πρέπει να αγωνίζονται για την ε, υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους ε, και για να μπορέσουν να ελέγξουν την σωστή διεξαγωγή των έργων. Στην περίπτωση αυτή είναι πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα διότι υπόθηκε πολύ σωστά ότι διαπιστώθηκε στην μελέτη επιπτώσεων ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες για την γειτονική χώρα Επί της αρχής λοιπόν δεν χρειάζεται να ε, ενημερώσει κανείς ε, την άλλη χώρα. Εάν λοιπόν εγώ θέλω να χτίσω κάτι και ε, διαπιστώσω ότι αυτό δεν θα ενοχλήσει το γείτονα, τότε δεν χρειάζεται να τον ενημερώσω. Νομίζω ότι είναι συνηθισμένο να μιλάει κανείς με τους ε, γείτονες του για τέτοια πράγματα. Έχουμε μία συζήτηση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, διότι το θέμα αυτό δεν το έχω καταλάβει πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει εδώ ένα κενό στον νόμο. Πρέπει πάντα να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης, ε, άσχετα το αν υπάρχει καλή συνεργασία ή όχι. Εξέτασα τα έγγραφα και η Τσεχία λέει ότι ενημερώθηκε το Βερολίνο. Εγώ δεν ε, βρίσκω τον παραλήπτη στο Βερολίνο. Οι Τσέχοι μπορεί απλά να έστειλαν μια απλή επιστολή, αλλά οι Γερμανοί δεν φαίνεται να έχουν λάβει κάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης ε, και ερωτώ μπορούμε να στείλουμε επιστολή στην Τσεχία να μας ε, πούν ποιον ενημέρωσαν από τη γερμανική πλευρά. Διότι οι Γερμανοί λένε ότι δεν γνωρίζουν τίποτα. Αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή αποδείξει σχετικά με την πληροφορία αυτή. Και δεύτερη παρατήρηση. Έγινε η σχετική έρευνα και ε, εφόσον διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αρνητικέ επιπτώσεις για τη Γερμανία, δεν έχουμε πρόσβαση στο σύνολο της νομοδότησης. Εγώ ούτως ή άλλως όχι, διότι τι είμαι, απλώς ευρωβουλευτής είμαι. Αλλά η Κομισιόν έχει πρόσβαση, μπορούμε να στήσουμε από την Τσεχία να αναγνώσουμε την ε, μελέτη. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά για τρεις λόγους. Καταρχάς θα ήθελα να γνωρίζω πώς ενημερώθηκε η γερμανική πλευρά. Δεύτερον, ε, δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην ε, γνωμοδότηση. Και διαπιστώνω ότι η Τσεχία έκανε την έρευνα που έπρεπε, διαπίστωσε ότι η γειτονική χώρα δεν ε, θα υποστεί αρνητικές συνέπειες. Πιστεύω ότι πρέπει να ξαναστείλουμε επιστολή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος διότι είναι σημαντικό πάντα να ενημερώνεται η γειτονική χώρα σε περίπτωση διασυνοριακών έργων. Όταν ε, χτίζει κανείς ένα σπίτι, ενημερώνει το γείτονα. Δεν ε, φτάνει να πω εγώ ότι δεν θα ενοχληθεί ο γείτονα. Αυτό λοιπόν ε, αποτελεί κενό νομοθετικό. Θα πρέπει να ορίσουμε σαφώς λοιπόν ποιες περιοχές θεωρούνται διασυνοριακές και να υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Και φυσικά όταν χτίζει κανείς πυρηνικό εργοστάσιο θα πρέπει να ενημερώσει το γείτονα. Και επίσης όταν έχουμε διασυνοριακούς οικότοπους ε, θα πρέπει να ε, συνεννοούμε με τον ε, γείτονα, αλλά σε περιπτώσεις άλλων μέτρων δεν προβλέπεται απαραίτητα κάτι τέτοιο. Και εάν η μελέτη επιπτώσεων δείχνει ότι δεν θα ενοχληθεί ο γείτονα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να τον ενημερώσω. Ανοιχτή λοιπόν να παραμείνει αυτή η αναφορά και θα θέλαμε να δούμε το σύνολο της ε, σχετικής νομοδότησης και να διαπιστώσουμε ποιος ήταν ο παραλήπτης ε, από την γερμανική πλευρά. Και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να φροντίσουμε να υπάρχει υποχρέωση αμοιβαίας ενημέρωσης στο πνεύμα καλής γειτονίας. και μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει αυτή η υποχρέωση να ισχύει διπλά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να πω κάτι για αυτά που είπε ο συνάδελφος. Η υποχρέωση θα πρέπει να είναι όχι μόνο υποχρέωση ενημέρωσης, διότι οι Τσέχοι λένε ότι ενημερώσαμε. Η υποχρέωση θα πρέπει να είναι για αποδεδειγμένη κοινοποίηση και από τις δύο πλευρές. Διότι αλλιώς θα λένε μένω ότι εμείς ενημερώσαμε, δε ότι δεν ενημερωθήκαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω, συνάδελφοι, ότι πρόκειται για μία αναφορά ηλικίας 4 ετών. Ήδη έχει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013. Είχαμε γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΝΒΗ. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει διαπιστώσει να υπάρχει παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Επιπλέον, η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, κατόπιν αιτήματος της ΕΝΒΗ κατέληξε ότι η σχετική οδηγία δεν θα οδηγούσε τις ε, τσεχικές αρχές να καταλήξουν σε διαφορετικό ε, συμπέρασμα από αυτό στο οποίο κατέληξαν το 2010. Η Κομισιόν λοιπόν διαπιστώνει ότι επισήμως δεν υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις παρότι μπορεί κάποιοι να νιώθουν ότι υπάρχουν. Εγώ κάποτε ζούσα δίπλα σε καμπαναριό. Στην αρχή πρόσεχα κάθε φορά που χτυπούσε, αλλά μετά από κάποιο διάστημα συνηθίζει κανείς. Μέσα, πιθανότατα στα τέσσερα αυτά χρόνια, να μην είναι πια τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Πίτερ, ε, έχω κατανόηση, αλλά από την άλλη θα ήθελα να κλείσουμε την ε, αναφορά αυτή. Είναι παλιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Έχουμε ε, προσπαθήσει να συλλέξουμε πληροφορίες από όλες τις πλευρές. Μπορώ να το κάνω αυτό. Πίτερ, έλα. Πάντα μου αρέσει να κλείνουμε αναφορές. Υπάρχουν όμως δύο προβλήματα. Πρώτον, ε, σωστά, πρέπει κάποια στιγμή να πει κανεί στον αναφέροντα ότι υπάρχουν ε, τρόποι διαδικαστική προσφυγή ε, και να ακολουθήσετε αυτήν, για παράδειγμα, σε περίπτωση που δεν έχω πρόσβαση στη γνωμοδότηση. Ο Τσέχος δικηγόρος μου, εάν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια, διότι αυτό δεν είναι διαφάνεια. Κατά τη γνώμη μου εδώ πέρα ε, έχουμε ένα κενό στη λογική του δικαίου. Εάν είναι εντάξει η γνωμοδότηση, τότε πράγματι οι τσεχικές αρχές ε, θα έχουν ενεργήσει σωστά. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που κάνανε και πιθανότατα να φταίει ο νόμος ε, και γι' αυτό παρακαλώ όταν έχουμε οικοδομικά έργα σε δυσνορικές περιοχές που δεν βρίσκονται σε οικοτόπους, όσον αφορά αυτά τα έργα θα πρέπει να αλλάξει το θέμα της υποχρέωσης κοινοποίησης και ενημέρωσης. Και επίσης ε, είναι δύσκολο να πούμε να ακολουθήσει τη δικαστική οδό όταν ε, δεν έχει πρόσβαση κανείς ε, στα σχετικά έγγραφα, στην ε, σχετική έκθεση. Υπόσχομαι όμως στην Πρόεδρο ότι εάν γίνουν όλα αυτά μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά, αλλά σήμερα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Διότι νομίζω ότι απαιτούνται κάποιες ενέργειες από εμάς στην Επιτροπή. Έχουμε δύο πράγματα ακόμα που πρέπει να ξεκαθαριστούν. Και ε, είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε του πολίτε. Αν δεν λαμβάνουμε τι πληροφορίες που πρέπει, τότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Πρόεδρος. Πείτε. Μπορώ να σου υπενθυμίσω πάλι ότι είναι τεσσάρων ετών η αναφορά αυτή και εσένα σου αρέσει να κλείνεις αναφορές όταν όλα έχουν γίνει. Τα πάντα έχουμε κάνει για την περίπτωση αυτή. Αυτό που θα μπορούσες να κάνει για να σε κάνω ακόμα πιο ευτυχή είναι να σου υποσχεθώ ότι θα κλείσουμε την αναφορά στέλνοντας ε, με εξαιρετικά ευγενική επιστολή στον αναφέροντα μαζί με τις νομικές πτυχές ε, που έδωσε η νομική υπηρεσία στην ΕΜΒΗ και να δώσουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε και θα υπογράψω καλλιγραφικά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Μπορούμε. Δεν έχει λογική να κάνουμε κάτι άλλο. Επιστολή προς την ΕΝΒΙ πρέπει να στείλουμε. Θα στείλω αντίγραφο της επιστολής στην ΕΝΒΙ αν αυτό είναι εντάξει. Κλείνουμε την αναφορά και δίνουμε όλες τις πληροφορίες στον αναφέροντα ενημερώνουμε και την Επιτροπή ΕΝΒΗ, της ε, κοινοποιούμε αυτήν την ε, επιστολή κλεισίματος της αναφόρας. Ωραία. Αυτά, καλό μεσημέρι, καλό γεύμα και τα λέμε στις 3.